Dear colleagues, like to ask you to take your seat and all the guys who don't want to join our meeting. Θα ήθελα να σας ζητήσω να καθίσετε και όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη σημερινή μας συνεδρίαση παρακαλώ να αποχωρήσουν γιατί πρέπει να αρχίσουμε. Ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης και η Επίτροπος Τάιζεν πρέπει να φύγουν οπότε πρέπει να αρχίσουμε αμέσως. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κανένα σχόλιο για την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Βάλτη Νομπρόφσκι, Αντιπρόεδρο και Επίτροπο για τον Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο και τη Μαριάν Τάιζεν, Επίτροπο για την Απασχόληση Κοινωνικέ Υποθέσει, Δεξιότητε και την Εργασιακή Κινητικότητα, που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μα για μια, για μια κοινή ε, συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Απασχόληση για να συζητήσουμε τα ε, κοινά αυτά θέματα. Ο κύριος Μοσκοβισή δεν μπορεί να είναι εδώ εξαιτία ε, ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας παρουσιάσει τα CSR που προκύπτουν από την αξιολόγηση της εθνικής μεταρρύθμισης ε, τις ειδικές στις τάσης, κάτι το οποίο θα συζητηθεί στο ΕΚΟΦΗΝ τον Ιούλιο. Αυτό το γεγονός που ολοκληρώνει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2016 είναι τμήμα του πλαισίου λογοδοσίας που αναφέρεται στη, στον κανονισμό για, για, για ε, τα, το πακέτο 6 μέτρων. Ε, θα ακούσουμε τους επιτρόπους και στη συνέχεια θα έχουμε ε, γύρους ερωταποκρίσεων. Να δώσω λοιπόν το λόγο καταρχάς στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ντομπρόφσκης. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ε, σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή. Ε, Από κοινού με την κυρία Τάιζεν, ώστε να σας παρουσιάσουμε τη συστάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομικές πολιτικές για τις επόμενους 12 με 18 μήνες. Υπάρχουν τρεις ε, πολιτικές προτεραιότητες, η ενίσχυση της επένδυσης, ε, η συνέχιση των διοικητικών ε, μεταρρυθμίσεων και οι υπεύθυνε δημοσιονομικές πολιτικές. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια καλύτερη ανάκαμψη, μείωση της ανεργίας, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θεμελίωση περαιτέρω ευημερίας. Και επίσης είναι μη, ε, επειδή θέλουμε να σταθεροποιήσουμε ακόμη περισσότερο την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, θέλουμε να ολοκληρώσουμε και τη Συμφωνία για την Τραπεζική Ένωση, αλλά είμαι ε, βέβαιος ότι μόλις ακούσατε περισσότερα για αυτό το θέμα από τον συνάδελφο που μόλις αποχώρησε. Να περάσουμε τώρα στις ειδικέ αναχώρα ε, ιδιαιτερότητες. Ε, υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες ε, που αντανακλούν τις προκλήσεις των διαφόρων κρατών μελών. Γι' αυτόν υπάρχουν όλο και περισσότερες λεπτομερείς συστάσεις για τις χώρες που αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις. Οι συστάσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τις ε, διάφορα στοιχεία που αφορούν και την Ευρωζώνη ε, και την ε, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Έχουμε λοιπόν μία έκθεση που αφορά ολόκληρη την Ευρωζώνη, όπως επίσης και την έκθεση, την έρευνα που αφορά την ανάπτυξη της Ευρωζώνης τα, την τελευταία χρονιά. Ε, οι συστάσεις αυτές ε, που αφορούν την Ευρωζώνη δημοσιεύονται ώστε να μπορούν να ε, ληφθούν υπόψη στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης στις πολιτικές τους. Όλες οι ειδικές αναχώρα συστάσεις έχουν, στοχεύουν συγκεκριμένα θέματα. 89 συστάσεις θα δημοσιεύσουμε πάνω από 150 είχαμε πριν από δύο χρόνια. Επομένω είναι πιο εστιασμένη η κατάσταση. Επίσης έχουμε ε, ιεραρχήσει τα πράγματα με έντονο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους ε, και τους εμπλεκόμενους φορείς των ενόγων χωρών. Επίσης έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να διαβουλευθούν ε, με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους όταν ε, ε, επεξεργάζονται έγγραφα που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο δημοκρατικό διάλογο σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε μία τακτική και πιο διαφανή ανταλλαγή απόψεων μαζί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, υπήρξαν συστηματικές επισκέψεις στα κράτη-μέλη και μπήκαμε σε ε, συζητήσεις με ε, βασικούς παίκτες στα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις προκλήσεις, τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις, όπως επίσης και τα περισσότερα εμπόδια στις μεταρρυθμίσεις αλλά και στις επενδύσεις. Είναι ε, συγκεκριμένο το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή, εφόσον βρισκόμαστε σε μία περίοδο ανάκαμψης, μειώνεται η ανεργία, αλλά παραμένει υψηλή σε αρκετές χώρες ε, και ιδιαίτερα η ανεργία μεταξύ των νέων και η μακροχρόνια ανεργία δημιουργεί ανησυχίες ε, ε, έχει προχωρήσει λοιπόν η δουλειά μας για την εξάλληψη των μακροοικονομικών ανισοτήτων, αλλά ακόμη έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ε, ε, η ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, όπως η νομισματική πολιτική, η οποία βοηθά στην ανάκαμψη, επειδή είναι χαμηλή η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, επίσης ε, οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών παρημένουν σε χαμηλά επίπεδο, κάτι το οποίο ε, είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καθαρό ε, εισαγωγέα. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα περιμένουν να συμβούν. Ε, ε, ενδεχομένως η αίσθηση του κατεπήγοντος να χάνεται σε μερικές περιπτώσεις. Κάποιες χώρες έχουν κάνει κάποια μικρή πρόοδο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιάς της συστάσεις αναχώρα και αυτό δεν είναι αρκετά καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, τη βελτίωση των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ε, και ε, των προβλημάτων κοινωνικής, κοινωνικών υποδομών και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες δεν θα υπάρχουν για πάντα. Σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή θα χρειαστούμε θα, ολοκληρωθεί αυτή η ευνοϊκή περίοδος ε, όπου η ανάπτυξη ε, επικουρείται, συνεπικουρείται από, ε, σημαντικές, από σημαντικούς παράγοντες. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις αδυναμίες των οικονομιών μας. Όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων έχουμε μία ε, προσέγγιση εκ των προτέρων ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα κάποιες πολιτικές. Προτείναμε λοιπόν benchmarking και ε, πολλαπλής συμμόρφωσης εξέτασης σε διάφορες περιπτώσεις γιατί χρειάζεται πολιτικό σθένος ε, η διοικητική μεταρρύθμιση. Κάποια έχουν και μια δημοσιονομική πτυχή, κάποιες δεν έχουν. Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά ε, την ε, διοικητική ε, υποδομή και γι' αυτό ακριβώς έχουμε μία Επιτροπή Υποστήριξης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και υπέβαλε μία πρόταση για ένα συγκεκριμένο μέσο το οποίο θα θα ε, διευκολύνει ακόμη περισσότερο τα κράτη-μέλη. Ε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και τη δική σας υποστήριξη για το πρόγραμμα αυτό. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης και αυτά ε, βοηθούν τα κράτη-μέλη στις μεταρρυθμίσεις στις οποίες θέλουν να προβούν και προσπαθούν να εφαρμόσουν τις συστάσεις. Να περάσω τώρα σε κάποιες από τις λεπτομέρειες συγκεκριμένων συστάσεων αναχώρα. Καταρχάς, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που διευκολύνει την επένδυση. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε εστίαση στην χαμηλή αποδοτικότητα, και στην έλλειψη διαφάνειας και αυτό ήταν ένα πρόσκομα στην ε, ε, ε, ανάπτυξη των επενδύσεων πρέπει να προσπαθήσουμε και να ενισχύσουμε το τραπεζικό μας τομέα και να ενθαρρύνουμε την, τις πιστοτικές μας υπηρεσίες, ε, επίσης συμμετοχή στην αγορά εργασίας ε, για να υπάρξει καλή ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ευελιξίας ε, στις, στην εργασιακή νομοθεσία, η διαβίου εκμάθηση και κατάρτιση, όπως επίσης και ο εξυγχρονισμός του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που πρέπει και από κοινωνικής και από οικονομικής ε, ε, απόψεω ε, να είναι βιώσιμα. Η κυρία Τάισεν θα σα πει περισσότερα ω προ αυτό. Και τρίτον, υπεύθυνε δημοσιονομικές πολιτικές σημαίνει ότι αυτές θα συνάδουν με το κοινό δημοσιονομικό μας πλαίσιο και με το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Επίσης ε, θέλουμε μια δημοσιονομική πολιτική που θα μας δώσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και περισσότερη ανάπτυξη. Πρέπει να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Πέρα από τις ε, συστάσεις ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαλε προτάσεις και στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών. Πρώτον, θα θέλαμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να ομαδοποιήσει ε, τρεις χώρες, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία ε, από ε, το από την ε, ομάδα στην οποία ανήκαν προηγουμένως και θεωρούμε ότι αυτή η διόρθωση είναι δυνατή. Επίσης, αξιολόγηση Βελγίου και Φινλανδίας. Ε, οι προσπάθειές μας βάσει του άρθρου 186 παράγραφος 3 που λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες ε, ε, θα ε, κρίναμε ότι είναι ε, μάλλον συμβατές. Όσον αφορά την Ιταλία, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες το 2017 και θα προβούμε τότε στην αξιολόγηση, στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Πορτογαλία και η Ισπανία δεν έχουν επιδιορθώσει το έλλειμμα τους σύμφωνα με το υπερβολικό χρέος. Έχουμε προτείνει Έχουμε κάνει προτάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ε, θα επανέλθουμε όμως στην κατάσταση για τις δύο αυτές χώρες ε, στις αρχές του Ιουλίου. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας ε, και υποθέτω ότι θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις κοινωνικές πτυχές η συνάδελφος κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ντομπρόφσκης. Κυρία Τάισεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Ο κόσμο τη εργασία αλλάζει ταχύτατα. Η ψηφιακή επανάσταση προσφέρει πολλέ ευκαιρίε, αλλά επιφέρει και σημαντικέ αλλαγέ και ιδίω για του απλού ανθρώπου. Οι αλλαγέ προκαλούν αβεβαιότητε και καμιά φορά ο κόσμο τα νιώθει χαμένα. Και είναι πραγματική ανησυχία για πολλούς που διαρωτώνται τι θα φέρει το μέλλον. Είναι λοιπόν αναγκαίο να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμιστικές μας προσπάθειες έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχουν στις ζωές των ανθρώπων και στις ευκαιρίες που τους ανοίγονται. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του φετινού χρόνου έχουμε βάλει την έμφαση στην ευκαμψία και στην ασφάλεια με κοινωνικό πρόσημο. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο προωθούμε και στα πλαίσια του Bill of Social Rights. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες έχουν αποφέρει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Οι συνθήκες της αγοράς εργασίας βελτιώνονται, η ανεργία μειώνεται, όμως χρειάζεται πολύ πολύ μεγαλύτερη πρόοδος. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε ακόμα 21 εκατομμύρια άτομα εκτός εργασίας, όταν γνωρίζουμε ότι έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια νέους άνεργους και ότι η φτώχεια έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος, χρειάζεται να φτιαχτεί ένα περιβάλλον φιλικό στην εργασία με τόνωση των ε, προσόντων με συμμετοχή, περισσότερη συμμετοχή των, Γερμανών, των, των γυναικών για το 2016 οι συστάσεις αναχώρα αναφέρονται στα θέματα αυτά. Ενθαρρύνουμε πολλές χώρες μέλη, Φιλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, να ενσωματίσουν καλύτερα κοινωνικά μέτρα, κοινωνικά μέτρα δραστηριοποίησης, κοινωνικά δίκτυα, με στόχο να επανέλθουν οι άνεργοι στις δουλειές, να ξαναβρούν δουλειά δηλαδή. Αυτό είναι σημαντική προτεραιότητα. Ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη να ενισχύσουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών. Αυτά ισχύουν και για χώρες όπως ε, η Γερμανία και η Ιρλανδία, επίσης για την φροντίδα των παιδιών, για τη Σλοβακία, για να δοθούν ευκαιρίες στις γυναίκες, να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, Γερμανία και Γαλλία. Πρέπει να μειώσουν τις ε, ε, διαφορές, τις ανισότητες δηλαδή στις αμοιβέ. Ενθαρρύνουμε ε, χώρες άλλες όπως η Ιταλία και η Βουλγαρία να εξασφαλίσουν δίχτυα ασφαλείας για όλους. Προωθούμε την ανάπτυξη προσόντων, την έκβαση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εργοδότες στην Ευρώπη που αναζητούν ειδικευμένου εργαζόμενους. Και οι εργαζόμενοι ψάχνουν να βρουν θέσεις δουλειά που να τα αποκλίνονται στα προσόντα τους. Πρέπει λοιπόν να φέρουμε αυτούς σε επαφή, βελτιώνοντας την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Έτσι όπως είπα, ώστε να ξαναβρούν δουλειά οι άνεργοι και να ανοίξουν περισσότερες προοπτικές για όλους. Η νέα ατζέντα για την Ευρώπη που θα σας ε, παρουσιάσουμε στην ολομέλειά σας, ανοίγουν αυτές τις δυνατότητες. Δεν γίνονται ειδικέ συστάσεις για τους μετανάστες για συγκεκριμένες χώρες, διότι οι βασικές χώρες υποδοχής στείλουν στα πόδια τους σημαντικές πολιτικές για την υποδοχή των ετούντων άσυλων και των μεταναστών. Προτείνουμε ωστόσο, κάνουμε κάποιες γενικές προτάσεις και συστάσεις για να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των ανθρώπων με μεταναστευτικό παρελθόν και ομάδες που αντιμετωπίζουν τριμενείς συνθήκες. Η νέα ατζέντα για, τα, για τις δεξιότητες δηλαδή περιλαμβάνει σχετικές συστάσεις και μέτρα. Αγαπητοί ευρωβουλευτές, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, εξαρτώνται από έναν ε, σοβαρό κοινωνικό διάλογο με συμμετοχή όλων των φορέων και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε διαφορετικά επίπεδα συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και στην διαχειρισμό των πολιτικών και στην εφαρμογή. Ορισμένες από τις πολιτικές ε, θα δούμε να συμμετέχουν, θα ζητήσουμε να συμμετάσχουν δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι στον κοινωνικό διάλογο και στους μηχανισμούς του. Και μια τελευταία λέξη, ε, λέξη συγγνώμη, για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει να εκμεταλλευτούν οι χώρες μέλη και να χρησιμοποιήσουν τα διαθροτικά ταμεία για να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους και να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις συστάσεις που κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, για να επιτύχουμε στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε την συμμετοχή όλων των διαφερονμένων μερών, των κυβερνήσεων, των κοινοβουλίων, το, της οργανωμένης κοινωνίας και βεβαίω του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω την πολύ θεμελιώδη συμμετοχή σας στην συζήτηση Αναμένω τις εκθέσεις σας και θα είδατε άλλωστε ότι οι εφετινές συστάσεις στοχεύουν σημαντικά σε ζητήματα κοινωνικά και απασχόλησης. Μόνο με την εξασφάλιση ότι αυτά θα ενταχθούν περισσότερο σε όλους τους ε, τομείς κοινωνικής πολιτικής θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια πραγματική κοινωνική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ Επίτροπε Τάισεν. Όπως σας είπα, ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης και η κυρία Τάισεν πρέπει να, βγουν, να φύγουν την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε έξι γύρους περίπου 15 λεπτών, έχουμε λοιπόν 90 λεπτά. Αυτή τη στιγμή μας μένουν 92 λεπτά. Οπότε σας παρακαλώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρούν το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι εισηγητές θα έχουν ε, από 3 λεπτά μετά 10 λεπτά για την απάντηση και για τους επόμενους 5 ε, γύρους, 4 εκ των οποίων θα διευθύνει ο αντιπρόεδρος Ουρσφοκ ε, της ΕΜΠΛ. Θα έχουμε 1,5 λεπτό για καθένα από τους συναδέλφους και συνολικά 10 λεπτά για τις απαντήσεις της Επιτροπής. Λοιπόν, πρώτος γύρος, οι εισηγητές. Πρώτος, Alfred Ζάντ τρία λεπτά και κατόπιν και κατόπιν Σοφία Ριβιέρα επίσης τρία λεπτά ο Άλφρεντ έχει το λόγο ευχαριστώ οι συστάσεις του 16 έγιναν με βάση το απλουστευμένο, εξορθολογισμένο εξάμεινο που ξεκίνησε το 2015 και τονίζουν περισσότερο τον στόχο και αφήνουν ε, τα μέτρα για την επίτευξή τους στις χώρες. Στα πλαίσια αυτά έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτη για τις επενδύσεις. Οι μακροοικονομικοί λόγοι έπαιξαν ε, το ρόλο τους για την έλλειψη επενδύσεων και ιδιωτικών και δημοσίων, για τη δημοσιονομική εξυγίανση και οι δημόσιες διοικήσεις προτιμούν ε, κοινωνικές και άλλες βράχοι δαπάνες. Μήπως θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα μακροοικονομικά εμπόδια και τα προβλήματα των ε, δημοσίων διοικήσεων. Γιατί όλα αυτά αποθαρρύνουν τις επενδύσεις, αλλά θα αρκέσουν, δεν νομίζω. Παρά το ΕΦΣΥ, παρά τα διευθυντικά ταμεία, η έλλειψη επενδύσεων και δημοσίων και ιδιωτικών ε, είναι κάτι βασικό πλέον στην ενιαία αγορά. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις λένε ότι πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις. Συμφωνείτε ότι χρειαζόμαστε νέες προτάσεις πολιτικής που θα βοηθήσουν να αυξηθούν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Επίσης, το 2016 οι συστάσεις για την απασχόληση και, την, ε, ε και τα κοινωνικά μέτρα είναι 114. Επειδή έχουμε λιγότερες ε, συστάσεις φέτος, είναι σαφές ότι τα θέματα απασχόλησης και τα κοινωνικά θέματα παίζουν ε, ιδιαίτερα ξέχοντα ρόλο για το εξάμεινο. Πολλές συστάσεις αφορούν ε, τις δεξιότητες ε, και την κατάρτιση. 16 κράτη-μέλη έλαβαν ε, συστάσεις στους τομείς αυτούς, από 14 πέρυσι. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά η τραγωδία είναι ότι οι στόχοι του 2020 για την φτώχεια, την μείωση της φτώχειας, δεν θα επιτευχθούν και η κατάσταση θα είναι χειρότερη από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα για τους στόχους αυτούς. Δεν θα έπρεπε λοιπόν η καταπολέμηση της φτώχειας να πάρει πλήρη προτεραιότητα όσον αφορά τη διατύπωση των συστάσεων, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε οριστικά τη φτώχεια. Και οι συστάσεις αυτές γίνονται τμήματα της ε, κουλτούρας μας για αντιμετώπιση των προβλημάτων οικονομικής πολιτικής. Με βάση την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μόνο 4% εφαρμογή των συστάσεων. Και για πολλές ε, συστάσεις ε, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ουσιαστικά. Πάνω από 50%. Τα αποτελέσματα αυτά μοιάζει να δείχνουν, μοιάζει να δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη δεν δεσμεύονται να τις εφαρμόσουν. Αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μου, στο ότι δεν συμμετέχουν επαρκώς στα εθνικά κοινοβούλια παρά τις προσπάθειες. Άρα, Άρα, τρίτη ερώτηση. Υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να αλλάξει αυτή η διαδικασία, ούτω ώστε να συμμετέχουν ε, πολύ περισσότερο και με πιο, με πιο ουσιώδη τρόπο τα εθνικά κοινοβούλια. Η Σοφία για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, ε, Αγαπητοί Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να υπάρχουν ε, πολλές ανισότητες. Και απόδειξη είναι η αναχώρα συστάσεις που συζητάμε εδώ. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανισότητες εκπονήσαμε τη νέα στρατηγική όπου θέλουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες διαφορετικές ε, μεταρρυθμίσεις και περισσότερη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Για το ΕΛΚ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προϋπόθεση για να υπάρξει η κοινωνική δικαιοσύνη και για να είναι ο πολίτης ε, στο κέντρο των πολιτικών μας χρειαζόμαστε υπεύθυνη οικονομική προσέγγιση. Η υπερχρέωση υποθηκεύει το μέλλον για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Η εξέλιξη, η ανάπτυξη της κοινωνίας χρειάζεται μια κοινωνική οικονομία της αγοράς που να είναι εξορροπημένη και από τις δύο αυτές πλευρές. Γι' αυτό αντιμετωπίσαμε τεράστιες προκλήσεις. Η κατάσταση στην Ελλάδα των ε, προσφύγων, η καταπολέμηση τρομοκρατίας, οι απειλές κατά της εσωτερικής ασφάλειας, η τραπεζική κρίση. Οι κρίσεις που προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση γενικότερα και πώς όλα αυτά θέτουν ένα αμφιβόλο το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζουμε ή να αντιμετωπίσουμε τον δεχόμενο να εφαρμόσουμε κυρώσει για τις χώρες που έκαναν τεράστιες θυσίε για να εξορροπήσουν τα δημοσιονομικά. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία. Συζητάμε για δέκατα ή και εκατοστά μιας μονάδας για το έλλειμμα, αντί να στοχεύσουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα ανάπτυξη που να είναι η πρωταρχική μας ε, ιδέα και μέλημα διότι δεν είναι δυνατόν μέσω κυρώσεων να επιτύχουμε ανάπτυξη. Μια χώρα η οποία έχει επενεθεί για τις προσπάθειες που έκανε για να κάνει μεταρρυθμίσεις να εφίσταται κυρώσεις. Επειδή ένας από, τα, ένας από τους ε, λόγους αυτής της ε, μη επίτευξης των στόχων είναι ε, λόγος που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει επαρκής αλληλεγγύη στην προσέγγιση μας. Οπότε ερωτήσεις. Η Κομισιόν θα προτείνει να επιβληθούν κυρώσεις στα κράτη-μέλη. Αν και πρόκειται από ό,τι έμαθα να αναβληθεί για τον Ιούλιο αυτή η απόφαση. Δεύτερον, εάν η αναβολή των κυρώσεων θα διαρκέσει ένα χρόνο. Θα το κάνετε για να δείτε τα αποτελέσματα του 17. Θα ήθελα να μου πείτε ποιους στόχους έχετε και με τι κριτήρια αποφασίσατε, θα αποφασίσετε ενδεχομένω αυτήν την αναβολή. Σήμερα συζητάμε αυτές τις συστάσεις, ενώ το ΕΚΟΦΗΝ τον Ιούλιο, από ό,τι φαίνεται, θα εγκρίνει την απόφασή του τον Ιούλιο, ενώ το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει τον Οκτώβριο. Οπότε όλη η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμείνου θα πρέπει να τροποποιηθεί για να μπορέσουμε να εισαγάγουμε περισσότερο δημοκρατία. Γι' αυτό προτείνω η Επιτροπή Απασχόληση να μπορέσει να υποβάλει έκθεση πρωτοβουλία όπω και η ΕΚΟΝ και να μην υποβάλει μόνο γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα παρακαλώ να σας ζητήσω να τηρήσετε το χρόνο σας, γιατί διαφορετικά οι τελευταίοι που θα πάρουν το λόγο δεν θα έχουν το λόγο, το, τη δυνατότητα να ε, θέσουν τις ερωτήσεις τους. Πρώτα ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Ντομπρόφσκης, για να απαντήσει. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. για το πρώτο ερώτημα όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τα προσκόμματα στις επενδύσεις. Πράγματι, φέτος ε, εστιάσαμε το, την προσπάθειά μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αλλά και τις συστάσεις μας όσον αφορά τα εμπόδια που υπάρχουν στις ε, επενδύσεις ε, λόγω της αποτελεσματικότητας της, των των, ε, διοικη, των διοικήσεων ε, ή διαφόρων συμφορήσεων που υπήρχαν ε, στη διαδικασία για τις επενδύσεις κλπ. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων βάσει των προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί όχι ως τώρα 100 δισεκατομμύρια ε, δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων έχουμε αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο δείχνει ότι το επενδυτικό πρόγραμμα για την Ευρώπη και η προσπάθεια ύπαρξης 350 δισεκατομμυρίων επιπλέον σε επενδύσεις έχει δρομολογηθεί. αυτό που τώρα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε περαιτέρω τις επενδύσεις ε, με νεότερα ε, μέσα ή με την επέκταση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για τις ε, επενδύσεις. Με ποιο τρόπο ακριβώς θα γίνει αυτό. Το αξιολογεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους ερχόμενους μήνες. Εν πάση περιπτώσει, η προτεραιότητα για τις επενδύσεις ε, εξακολουθεί να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα, κάποιοι αναφέρατε ε, αυτό που είπα και εγώ ότι όντως υπάρχει γενικότερα μεγαλύτερη πρόοδος, αλλά η πρόοδος δεν είναι επαρκής και ότι γι' αυτό ε, πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας για να βελτιώσουμε την εφαρμογή των συστάσεων. Αλλά όπως κάθε φορά τονίζω, οι συστάσεις αυτές δεν είναι διαταγές. Δεν υπάρχει μηχανισμός ε, επιβολής της εφαρμογής ε, των συστάσεων αυτών αναχώρα. Επομένως, η βελτίωση της εφαρμογής πιστεύουμε ότι περνάει από τη βελτίωση της ε, κυριότητας, μεγαλύτερης δέσμευσης ε, των κυβερνήσεων ε, των κοινωνικών εταίρων και άλλων εμπλεκομένων φορέων, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, να εντοπιστούν οι προκλήσεις πολιτικής και να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές. Επίσης, Προφανώς υπάρχουν κάποια μέσα υποστήριξης των κρατών μελών για την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα μέσω τεχνικής υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αναφέρθηκα και στην, στο πρόγραμμα υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Προσπαθούμε λοιπόν να ενισχύσουμε τα εθνικά κοινοβούλια προ αυτή την κατεύθυνση και αυτό αποτελεί επίση προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, ως προς το, τα ερωτήματα που είχαν να κάνουν ε, με την ε, εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τις ενδεχόμενες ε, κυρώσεις. Ως πώς γνωρίζετε, οι αποφάσεις για τη διαδικασία υπερβολικού λιματος βάσει του άρθρου 126 της συνθήκης στην περίπτωση της Πορτογαλίας και της Ισπανίας έχει αναβληθεί Μέχρι τον Ιούλιο δεν ε, υπάρχουν άλλα σχέδια αναβολής, περαιτέρω αναβολής των συγκεκριμένων αποφάσεων. Εγώ δεν μπορώ να προκαταβάλω τα, ε, τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τον Ιούλιο. Αλλά ως θεματοφύλακα των συνθήκων έχουμε καθήκον ε, να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το πρώτο βήμα είναι η επίσπευση της διαδικασίας ε, του υπερβολικού ελλείμματος και αυτή τη στιγμή έχει εγκριθεί αυτό ε, στο ε, Συμβούλιο, τότε θα γίνουν περαιτέρω βήματα. Είναι δυνατόν να γίνουν περαιτέρω βήματα. Βεβαίως ε, εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος ε, την ε, προσπάθεια μεταρρυθμίσεων και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και επέτρεψε στι χώρε αυτές να επιστρέψουν σε πορεία ανάπτυξη, αλλά πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει το γεγονός ότι όλες οι χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν την οικονομική τους ανάκαμψη και θετικό οικονομικό περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι που σε κάθε περίπτωση πρέπει να λάβει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αποφασίζει τα επόμενα βήματα σε σχέση με τη διαδικασία αυτή ε, υπερβολικού ελλείμματος. Η κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στα Ολλανδικά αν μου επιτρέπετε. Η φτώχεια είναι πράγματι, η καταπολέμησή της δηλαδή, ένα, μια από τις προκλήσεις που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και γνωρίζουμε ήδη ότι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο, δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε την φτώχεια στο ποσοστό που θα θέλαμε. Θα τη διατηρήσουμε στο ε, σημερινό επίπεδο, αλλά δεν χρειάζεται να μειώσουμε τους στόχους μας. Εξακολουθεί πάντως να αποτελεί προτεραιότητά μας σε ό,τι αφορά τις ειδικέ αναχώρας συστάσεις για το 2016 θα δείτε ότι περίπου οι μισές από τις χώρες μέλη λαμβάνουν συστάσεις που αφορούν και θα επιδράσουν στα επίπεδα της φτώχειας στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι δύσκολο βέβαια να γίνει μια σύγκριση ανάμεσα σε φτώχεια και ένα διαμάντι, αλλά με την έννοια ότι είναι πολυδιάστατη η φτώχεια. Έχει πολλέ δηλαδή, πλευρέ, όπω ακριβώ έχει ένα διαμάντι. Με αυτήν την έννοια προσπαθώ να πω ότι χρειάζεται προσέγγιση από πολλέ πλευρέ. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στι συστάσει μα, καταδείχνοντα στι χώρε μέλη που πρέπει να αναλυφθεί εργασία. Για να πρέπει να γίνει δουλειά δηλαδή. Και στα επιδόματα ανεργίας και στην κοινωνική προστασία και ταυτόχρονα να ληφθούν και μέτρα δραστηριοποίησης διότι όσο γρηγορότερα βγει και ο καλύτερος μάλλον τρόπος για να βγει γρηγορότερα από τη φτώχεια κάποιος είναι να βρει δουλειά. Κάνουμε συστάσεις, ειδικές συστάσεις και για τα παιδιά. Αν θέλουμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της φτώχειας πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωση των πολύ νέων παιδιών και κάνουμε συστάσεις για αυτά. Ζητούμε δηλαδή καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας για την φροντίδα των παιδιών και επίσης ορθή κατάρτιση, καλή εκπαίδευση των παιδιών από την πολύ νεαρή ηλικία. Ασχολούμεθα και με την μακρόχρονη ανεργία. Επίσης, ε, σημαντικό πεδίο αγώνα κατά της φτώχειας. Σε πολλές χώρες κάνουμε συστάσεις να θεσπίσουν ένα ελάχιστο μισθό ή να αυξήσουν τον ήδη υπάρχοντα ελάχιστο μισθό. Κάνουμε λοιπόν σχετικές συστάσεις. Ορισμένες χώρες ε, μέλη μπορούν να υποφεληθούν από τα διαστατικά ταμεία για αυτά. Μιλούμε επίσης και για αυτή την ε, σφήνα, τη φορολογική σφήνα, την επιβάρυνση δηλαδή με φόρους της εργασίας, που καμιά φορά χτυπάει και την εργασία τη χαμηλότερα αμοιβόμενη εργασία και τα χαμηλότερα, δηλαδή χαμηλότερου εισοδήματο νοικοκυριά. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους που έχουν χαμηλότερα προσόντα και δεξιότητες να είναι και το πιθανότερο είτε να παραμείνουν είτε να ε, ε, μπουν στη φτώχεια. Έτσι λοιπόν χρειάζεται η προσέγγιση, προσέγγιση της φτώχειας από πολλές πλευρές. Και αυτή είναι μια διαρκή ανησυχία μα και αυτήν υποδεικνύουμε στι διάφορε χώρες μέλη με την έννοια ότι πρέπει να περιλάβουν στι ατζέντε του συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει. Αν θέλουμε κοινωνική Ευρώπη πρέπει να βοηθήσουμε του στοχότερους να βγουν από τη φτώχεια. Ευχαριστώ. Δεύτερο γύρο, τέσσερις ομιλητέ από πλευράς μας. Ενάμιση λεπτό ο καθένας παρακαλώ. Θα υπάρχει ένα αλλαγή ομιλητών Έκον και Έμπλε. Ντάριο Ροζάτη, ΕΛΚ από την Έκον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση για τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόσκης. Ε, Καλώ ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε. Μία από τις αδυναμίες ε, της ε, παρούση ανάκαμψης στην Ένωση είναι η πολύ αργή άνοδος τη παραγωγικότητα. Είναι μισό από ό,τι ήταν την περίοδο 2000-2008 και λιγότερο από ένα τρίτο από ό,τι ήταν στις δεκαετίες του 80 και του 90. Αυτός είναι ο βασικός παράγον που ε, εξηγεί το χαμηλό βαθμό ανάπτυξης. Ε, πώς την εξηγείτε εσείς και τι συστάσεις ε, προτίθεται να απευθύνει η Επιτροπή στα κράτη-μέλη για να διορθωθεί το θέμα αυτό. Δεύτερη ερώτηση προς την Επίτροπο Τάισιν. Το φετινό ευρωπαϊκό εξάμεινο εστιάζει περισσότερο στην ανεργία και την κοινωνική απόδοση οι αποφάσει που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριληφθούν άλλοι τρει δείκτε για την απασχόληση στον πίνακα αποτελεσμάτων, υποτίθεται ότι θα διεύρυνε το πεδίο εφαρμογή τη ανάλυση και θα την έκανε πιο συνολική. Πώ αντανακλάται αυτό στι αναχώρα συστάσει, και ποιε είναι οι συγκεκριμένε συστάσει προ τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η κατάσταση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και συγκεκριμένα αντιμετωπίζουν και την ε, νομοθεσία που προστατεύει την απασχόληση στα κράτη-μέλη. Και να ορίστε. Δωρεάν σας δίνω και πέντε δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ, Ντάριου. Σοσιαλιστές τώρα, έμπλα. Η Μαρία Ζουάου Γουντρίγιους. Ευχαριστώ πολύ για τα πέντε δευτερόλεπτα, λέει η κυρία Μαρία Ζουάου Γουντρίγιους. Καταλαβαίνουμε ότι κατά το παρόν ευρωπαϊκό εξάμεινο μετά από τις ε, έντονες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου, διαπιστώνουμε ότι λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η κοινωνική διάσταση. Αλλά κατά τη γνώμη μας εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Διότι αν πραγματικά θέλουμε να μειωθεί η υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε βελτίωση των κοινωνικών δικτών παντού στην Ευρώπη και να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες πρέπει να έχουμε πιο φιλόδοξη στρατηγική. Πρώτον, πώς ορίζουμε τους στόχους. Οι στόχοι πρέπει να αφορούν την ανεργία, τις κοινωνικές ανισότητες και τα κοινωνικά πρότυπα. Κατόπιν, πώς σχεδιάζονται οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να σχεδιάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα. Τρίτον, υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν κοινωνικές επενδύσεις εντός του γενικού πλαισίου επενδύσεων. Και τέταρτον, ο ρυθμό δημοσιονομικής εξυγίανση δεν θα βαθύνει τις κοινωνικές ανισότητες και δεν θα υπονομεύσει την εγχώρια ζήτηση. Και πρέπει να βρούμε τρόπο να μειώσουμε τις μακροοικονομικές ανισότητες. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι όλες οι χώρες πρέπει να συμβάλλουν. Οι λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες δεν θα πρέπει να κάνουν εσωτερική υποτίμηση, θα πρέπει να μπορέσουν να επενδύσουν και να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Αλλά και οι χώρες με υψηλή ανταγωνιστικότητα πρέπει να επεκτείνουν, να βελτιώσουν την εσωτερική του ζήτηση. Αυτή η στρατηγική δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να ολοκληρωθεί ή ο ναι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος, Γιώχιμ Σταμπάτη. Αλλά θα μιλήσει και από πλευρά των δύο επιτροπών, οπότε έχει τρία λεπτά. Μία παρατήρηση σε αυτά που είπε ο Επίτροπος Ντομπρόσκης. Πολύ συχνά και στο Κοινοβούλιο και στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές ακούω ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη, επενδύσεις, έχουμε πολύ ψηλή ανεργία, κάτι έχουμε κάνει αλλά όχι επαρκή. Υπενθυμίζω αυτό που είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ, ότι πρέπει να κάνουμε έντιμες προσπάθειες. Να δούμε τι γίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βαδίζει και πάλι προς τον κρεμό. Και αυτό έχει να κάνει με αυτά που έχει υποστεί από την Ευρωζώνη. Εδώ και τόσα χρόνια μας λένε ότι είναι εντελώς μη ανταγωνιστική η οικονομία της Ελλάδας. Και αν τους δώσουμε λεφτά δεν τους βοηθάμε αυτούς, αλλά τους πιστωτές τους. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Το θέμα είναι η επιβίωση της Ευρωζώνης, γιατί φοβόμαστε ότι εάν αποχωρήσει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη θα πάνε και άλλοι. Δηλαδή τι θα βοηθούσε πραγματικά την Ελλάδα. Την Ελλάδα θα τη βοηθούσε εάν αλλάξει η ε, ισοτιμία δεν αρκούν οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Δεύτερον, η Ελλάδα χρειάζεται πολύ έντονη περικοπή του χρέους τους και χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό χρηματοδότηση για να της δώσει μια όθηση, για να είναι σε θέση να βρουν δουλειά στη χώρα τους οι πολίτες και να μην χρειαστεί να μεταναστεύουν. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα για την αγορά εργασίας. Ο Υπουργό Οικονομικών της Ιταλίας είπε ότι αν αξιοποιήσουμε, εάν δεν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε των, ε, τις ε, αλλαγές για να υπάρξει ισορρόπηση, τότε πρέπει να αλλάξει η αγορά εργασίας. Και αυτό είναι το σκληρότερο μέτρο που μπορούμε να λάβουμε. Να συγκρίνω την Ελβετία με την Πορτογαλία. Όπω ξέρετε έχει υπάρξει μεγάλη ανατίμηση του ελβετικού φράγκου σε σχέση με το ευρώ. Τι έκαναν. Αύξησαν ε, πάρα πολύ τι ώρε εργασία χωρί να αυξηθεί το, χωρίς να αυξηθούν οι αποδοχές. Αυτή είναι μια εσωτερική υποτίμηση για να αντιμετωπίσουν την ανατίμηση του φράγκου. Τι έγινε στην Πορτογαλία αντίστροφα. Στην Πορτογαλία ο χρόνος εργασίας ε, πήγε από 38 σε 35 ώρες. Ποιες είναι οι επιπτώσεις. Η παραγωγικότητα μειώνεται. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Πορτογαλίας επίσης μειώνεται. Αλλά η Πορτογαλία πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Πρέπει να κάνει λοιπόν εσωτερική υποτίμηση. Πώς είναι δυνατόν ε, σε ένα τέτοιο πλαίσιο να επιτύχουμε τους στόχους μας αυτούς που όλοι θέλουμε. Ανάπτυξη, παραγωγικότητα, μείωση της ανεργίας, μείωση της ανεργίας των νέων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Επιτροπή. Πρώτα ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, για το ερώτημα ε, χαμηλής ε, ανάπτυξης της παραγωγικότητας. Όπως είπατε κι εσείς ε, ότι είναι αυτό που ευθύνεται για την χαμηλή οικονομική μας ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ο πρώτος ε, παράγοντας, ε, και είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, είναι η έλλειψη επενδύσεων. Γιατί στις, ε, με, τις επενδύσεις, τη μείωση των επενδύσεων μειώνεται η μελλοντική, το μελλοντικό δυναμικό ανάπτυξης και επίσης μειώνεται και το ποσοστό ανάπτυξης ο ρυθμός ανάπτυξης. Επίσης υπήρξαν και κάποιες μελέτες ε, από τον ΩΣΑ για την ε, αποδοτικότητα των αγορών, στις οποίες αναφερόταν ότι υπάρχει σοβαρή διαφορά μεταξύ ε, παραγωγικότητας από επιχειρήσει σε επιχείρηση. Υπάρχουν επιχειρήσεις των οποίων η χαμηλή παραγωγικότητα μένει εντός της αγοράς και ε, υπάρχει και μία χαμηλή ε, ανάπτυξη εξ αυτού. Υπάρχει λοιπόν μία σχέση. Αν θέλουμε μία ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και αν θέλουμε να επιτύχουμε υψηλά ποσοστά ευημερία, πρέπει να έχουμε και υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Αυτό ε, είναι και πίσω από τη λογική της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν ε, προτείνει να υπάρχει ένα ε, Συμβούλιο Εθνικής Ανταγωνιστικότητας ώστε να υπάρξει ανεξάρτητη, ανεξάρτητες συμβουλές επί πολιτικής προς τις χώρες είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή συζητιέται στο Συμβούλιο και ελπίζω ότι στο ΕΚΟΦΗΝ του Ιουνίου θα υπάρξει σύντομα μια απόφαση επ' αυτού. Όσον αφορά τώρα την καλύτερη ενσωμάτωση των κοινωνικών πτυχών στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Σας ευχαριστώ πολύ για την αναγνώριση της εργασίας που έχει ήδη λάβει η χώρα και συνεχίζει βέβαια αυτή ε, η εργασία, αλλά ε, η κυρία Τάισεν θα ε, πει περισσότερα από αυτού. Υπάρχει το ερώτημα επίσης για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Αναφερθήκατε και στη δημοσιονομική εξυγίανση δεν είμαστε πλέον ε, σε θέση συνολικής δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ε, είχα πει ότι σε γενικές γραμμές ε, στην Ευρωζώνη οι τάσεις είναι μάλλον αυξητικές. Εξακολουθούν να υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν ε, ονομαστικές, ε, υπάρχει μια ονομαστική μείωση και ε, η πραγματική μείωση, η πραγματική ανάπτυξη επίσης έχει αρχίσει να δρομολογείται. Ελπίζουμε συνολικά ότι μέσω των χαρτών πορείας κατά τους ερχόμενους μήνες θα επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαβουλεύσεων, ελπίζω ότι ε, θα περάσουμε σύντομα στην, στο, στο στάδιο 2. Για το ερώτημα που αφορά ε, την κατάσταση στην Ελλάδα. Όσον αφορά στην Ελλάδα, ε, ολοκληρώνουμε αυτή τη στιγμή μια πρώτη μας αναθεώρηση, αξιολόγηση ώστε να αξιολογήσουμε και την επόμενη, επόμενη δόση. Ε, ε, έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις κατά την τελευταία χρονιά και έχουν βοηθήσει στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ε, υπάρχει πάλι οικονομική σταθερότητα, υπάρχει μπορούμε να, να περιμένουμε ότι και η Ελλάδα θα επιστρέψει σε μία πορεία ανάπτυξης. Ε, ήδη 27 από τις 28 χώρες ε, της Ένωσης σημειώνουν οικονομική ανάπτυξη ε, και ελπίζουμε ότι και η Ελλάδα θα επιστρέψει ε, σε αυτήν την πορεία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά τώρα την ε, ε, εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Προφανώς δεν μπορείς να υποτιμήσει το νόμισμά σου όταν συμμετέχεις στο ευρώ. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο νομισματικής πολιτικής. Υπάρχουν βεβαίω. Ε, Υπάρχουν βέβαια ε, από νωρίς κάποιες ε, ε, πολιτικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα μετά. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μέσω της διαδικασίας μακροχρόνιων, μακροοικονομικών ανισοτήτων να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω, το λόγο στην, πριν την προεδρία στην κυρία και να δώσω το λόγο στην κυρία Τάισεν για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Ρωσάτη για το τι κάναμε με τους κοινωνικούς δείκτες ε, τους χρησιμοποιήσαμε ε, στις εκθέσεις για τις χώρες, ε, γιατί επέτρεψαν μια καλύτερη κατανόηση της κατάστασης ε, στις εν λόγω χώρες και εμέσως αντανακλώνται στις ανασύσταση εκθέσεις όσον αφορά την μακροπρόθεσμη ανεργία, τη μακροχρόνια ανεργία, την ανεργία των νέων. Ως προς αυτά βοήθησαν πολύ ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες συστάσεις. Όσον αφορά το ποσοστό ε, ε, ενεργού ε, συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ενεργού συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Έχουμε πολλές φορές τονίσει τη σημασία συμμετοχής της κοινωνικής προστασίας με την κινητοποίηση των ανθρώπων που χρειάζονται τέτοιου είδους προστασία. Όσον αφορά την ενεργεία των νέων, υπάρχουν κάποιες συστάσεις, λιγότερες από αυτές που αναμέναμε, γιατί ακριβώς υπάρχουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και με την βοήθεια, με την βοήθεια της διευκόλυνσης για τους νέους θα δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να συνεχίσουμε με αυτή την προσπάθεια. Αλλά φαίνεται και στις ε, αναχώρα ε, συστάσεις ε, Νομίζω ότι έξι κράτη-μέλη για τα οποία εκτός από την μακροχρόνια στρατηγική έχουμε προσθέσει και ειδικές συστάσεις ε, για ε, ένα στα τέσσερα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα την ε, απασχόληση και τις συμβάσεις απασχόλησης, εκεί έγιναν κάποιες παρατηρήσεις από τα κράτη-μέλη όσον αφορά το διτό χαρακτήρα της αγοράς εργασίας από ανεπίσημες συμβάσεις εργασίας σε πραγματικές συμβάσεις εργασίας, αλλά πρέπει να εξετάσουμε συγκεκριμένα είδη ε, συμβάσεων, γιατί ε, πρέπει να δούμε και τα, τις συμβάσεις αστικού δικαίου, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που αποκαλούνται αυτοαπασχολούμενοι, οπότε και εδώ υπάρχει ε, μια, ε, ε, ένας, μια διπλή μια δυτή κατάσταση στην αγορά εργασίας. Στην ερώτηση του κυρίου Ροντρίγκε όσον αφορά την ανισότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι στο τρίγωνο ε, δημοσιονομικής υπευθύνης υπευθυνότητας, ε, ε, σταθερότητα και επιπλέον επενδύσεις. Ε, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και φυσικά περισσότερη ευημερία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν συμβαίνει εν μια ανοιχτή, χρειάζεται χρόνο. Πιστεύουμε όμως ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλα αυτά τα μέτωπα μπορεί να επιφέρουν αποτελέσματα και όπως είπε και ο Βάλτης, με την εμβάθυνση της νομικής Νομισματικής Ένωσης θέλουμε περισσότερη ε, σταθερότητα. Ε, χρειαζόμαστε τη σταθερότητα ε, και για την Ένωση, για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αλλά και για να επιτύχουμε την φιλοδοξία που ανέφερε ο κύριος Γιούγκερ, ότι θέλουμε σύγκληση προς τα πάνω. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας και ας προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε για να το επιτύχουμε αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Ζήμων που προεδρεύσατε στο πρώτο τμήμα αυτής της ανταλλαγής απόψεων. Να δώσω το λόγο στον Νίλ Στούρβαλτς τώρα. 90 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους επιτρόπους για την παρουσία τους. Νομίζω ότι υπάρχει μια ε, θρησκευτική δογματική προσήλωση στην ιδέα της συνοχής και της σύγκλησης. Μια με, πανεπιστημιακή μελέτη Απέδειξε αυτό που δείχνουν και πολλές άλλες μελέτες, ότι δηλαδή η σύγκληση δεν επιτυχάνεται. Όσοι έχουν καλή μνήμη και τους αρέσουν οι ιστορικές ηρωνίες θα θυμούνται ότι ο Γκρέκορ Μέντελς έκανε την περίφημη μελέτη του της βοτανικής με τίτλο ε, «Πειράματα για υβριδικά φυτά». Τι κάνουμε λοιπόν εμείς τώρα. Έχουμε αυτή την ε, θρησκευτική προσήλωση και προσπαθούμε να κάνουμε πειράματα για υβριδικά κράτη. Και στην περίπτωση των παιδιών κάνουμε ε, πειράματα για υβριδικά παιδιά. Θα πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά. Ευχαριστώ. Ενρίκε Κάλβετ Σαμπόν, 90 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε να δούμε αν θα προλάβω να πω αρκετά πράγματα. Πρώτον, η διακυβέρνηση. Όλα αυτά είναι θέματα διακυβέρνησης. Όμως ε, πρέπει να πούμε ότι αν δεν είναι ρεαλιστική η διακυβέρνηση και εξαρτάται από μικροπολιτικούς ε, σκοπούς τότε δεν επιτυγχάνουμε τίποτα. Ε, αυτό το σύστημα για παράδειγμα προστήμων ε, πρέπει να αναθεωρηθεί, αλλά τουλάχιστον πρέπει να έχουμε κανόνε, Αλλά παρακαλώ να παρατηρείτε και τι δομέ και την διακυβέρνηση των χωρών. Για τι ορισμένε χώρε ε, δεν υπάρχει ε, ε καμία δυνατότητα πλέον ουσιώδου διακυβέρνηση. Και είναι διαφορετικό το πρόβλημα. Όπω καταλαβαίνετε, μιλάω για τη δική μου χώρα. Επιπλέον, πώ είναι δυνατόν, ίσω είναι και καλή αλλά πώ είναι δυνατόν να υπάρχουν λιγότερε συστάσει από πριν, από πέρυσι δηλαδή, για θέματα ανεργία των νέων. Ξέρω ότι η ανεργία των νέων ε, έχει αρχίσει κάπως να βελτιώνεται, αλλά πώς είναι δυνατόν να έχουμε λιγότερες συστάσεις. Τέταρτον, η ε, ελαστική ασφάλεια που λέμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι όποιος ε, είναι άνεργος βοηθιέται από την κοινωνία και αυτό σημαίνει πολλές δημόσιες δαπάνες. Να λαμβάνετε υπόψη λοιπόν και αυτό το θέμα. Και κάτι ακόμη για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης. Αυτό που λείπει είναι πρώτον να συνεχιστούν οι προσπάθειες για κινητικότητα μέσω και μιας κοινή γλώσσας και επίσης πρέπει να δούμε εναλλακτικέ λύσεις για τη δυναμική των ανισοτήτων που δημιουργεί προβλήματα και για την οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Μαρίσα Ματίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης. Νομίζω ότι δεν απαντήσατε στην ερώτηση που ετέθη για τις κυρώσεις, οπότε επανέρχομαι. Είπατε ότι η Επιτροπή πρέπει να εγγυηθεί ένα θετικό οικονομικό πλαίσιο, αλλά δεν απαντάτε συγκεκριμένα στις ερωτήσεις. Είναι δυνατόν, κατά τη γνώμη σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταχειρίζεται διαφορετικά χώρες που έχουν υπερβολικά ελλείμματα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται να συζητήσει κυρώσεις για Πορτογαλία και Ισπανία, αλλά όχι για το Βέλιο και τη Γαλλία. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ε, πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να φανταστώ είναι ότι Είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες προτιμήσεις για κάποιες κυβερνήσεις γιατί έχουν κάποια πολιτική φύση ή ότι η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη το οικονομικό βάρος των χωρών. Διότι αν θέλετε θετικό οικονομικό κλίμα όπως είπατε δεν καταλαβαίνω πώς να τον έχετε τέτοια συμπεριφορά. Και παρακαλώ απαντήστε επιτέλους για αυτό το θέμα των κυρώσεων. Και επιπλέον, αν θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι για το ε, πώς θα μπορούσε να επιβιώσει το ευρωπαϊκό όραμα και εγχείρημα με τέτοια ε, πολιτική. ο Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ πολύ. Η πραγματικότητα δείχνει ποιο είναι το αποτέλεσμα των οικονομικών πολιτικών σε μια ένωση δύο ταχυτήτων. Σε ορισμένους κάνουν ειδικέ ρυθμίσεις, ενώ άλλους τους εκβιάζουν, όπως στην Πορτογαλία η επίθεση στην κρατική κυριαρχία, η αιμονή σε διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, οι πολιτικές λιτότητας και τα σύμφωνα, οι επιθέσεις των χωρών που υφίστανται τρόικα οδήγησαν σε 25 εκατομμύρια φτωχούς. Η αύξηση των ανισοτήτων, η ανεργία, η επισφάλεια, οι επιθέσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η καταστροφή και η ιδιωτικοποίηση των ε, ε, δημοσίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην υγεία. Όλα αυτά οδηγούν σε έλλειψη ανάπτυξη και σε μείωση τη κατανάλωση. Μέχρι πότε θα συνεχίσει να επιμένει η Κομισιόν στην εφαρμογή τέτοιων πολιτικών μέσω των συστάσεων αναχώρα. Επιπλέον, από απαράδεκτε και αντιδημοκρατικέ, αυτέ οι συστάσει αυξάνουν τον αποκλεισμό σε χώρε όπω η Πορτογαλία. Παρά το ότι επιτύχαμε του στόχου για το έλλειμμα που μα έθεσε η Τρόικα, επιμένουν ακόμη περισσότερο το κρατικό έλλειμμα τελικά απορρόφησε το ιδιωτικό έλλειμμα και τώρα το κράτος ε, έχει δε, ε, ε, δισεκατομμυρίων. Κάτι που δεν επιτρέπει πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι δυνατόν να μας επιτρέψετε αναδιαπραγμάτευση για τις προθεσμίες και τα επιτόκια του δημοσίου χρέους. Ευχαριστώ Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση. Για τη σύγκληση. Όντως. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε σύγκληση με καλό ρυθμό πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση. Έκτοτε δυστυχώς ε, διεκόπη. Γι' αυτό προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι να επανεκκινήσει η διαδικασία σύγκλησης. Και όπως είπα, πρέπει να υπάρχει σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών, αλλά πρέπει να υπάρξει και εντός των κρατών μελών, δηλαδή μείωση των ε, εισοδηματικών ανισοτήτων. Και υπάρχουν τρόποι για να προωθήσουμε αυτή τη σύγκληση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμάει την ε, προσέγγιση ανταλλαγής ε, βελτίστων πρακτικών, καθορισμού προτύπων και προδιαγραφών, ούτω ώστε να προωθήσουμε το στόχο της σύγκλησης. Ε, τώρα, έχουμε ερωτήσεις για την διακυβέρνηση, γιατί έχουμε λιγότερες συστάσεις για την ανεργία των νέων, για την ευελικτοασφάλεια, flex security. Στο παρόν ευρωπαϊκό εξάμεινο μας ρωτάτε γιατί τα κάνουμε αυτά. Προτείνουμε λιγότερες αναχώρα συστάσεις, αλλά πιο στοχευμένες. Αυτό εκτιμήθηκε θετικά και σε έγγραφα του Κοινοβουλίου. Και αυτό σημαίνει ότι καταλάβαμε ότι αν όλα είναι προτεραιότητα, δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα. Πρέπει να επιλέξουμε προσεκτικά τι συστάσει κάνουμε και σε ποιου τομεί πολιτική τι κάνουμε. Αλλά τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα απασχόλησης και οι δείκτε επ' αυτών είναι πιο προβεβλημένα στην παρούσα διαδικασία και κατά πολέμη της ανεργίας είναι από τις βασικές προτεραιότητες. Και η Κομισιόν μία από τις πρώτες προτάσεις που έκανε αυτή η παρούσα Κομισιόν ήταν πώς θα επιταχύνουμε την ε, πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων και το σύστημα εγγύσεων για την ανεργία των νέων. Τώρα, πώς εφαρμόζεται το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω ότι ως θεματοφύλαξη των συνθήκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει το σύμφωνο αυτό. Η Επιτροπή αποφάσισε να ξαναδεί τα θέματα 126 της συνθήκης για την περίπτωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας αρχές Ιουλίου. Σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να προκαταλάβω τι απόφαση θα πάρει στις αρχές Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα περισσότερα για αυτό το θέμα. Για το θέμα σύγκρισης Γαλλίας και Πορτογαλίας και αν ε, εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ανάλογα με το κράτος μέλος και φυσικά αυτό είναι πολύ σοβαρό. Όπως τόνισε επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμόζουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με βάση κανόνες και με βάση τα στοιχεία. Λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική και νομική διακριτική ικανότητα που τις παρέχουν οι συνθήκες. Συγκεκριμένα για τη Γαλλία. Η Γαλλία πρέπει να διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμα του χρόνου, δηλαδή να είναι κάτω του 3% του ΑΕΠ του χρόνου και η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση. Και Ελπίζουμε να μας υποβάλει το πρόγραμμά της η Γαλλία γι' αυτό. Για το Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς κυρία Τάισεν, θα είμαι σύντομη, θα προσπαθήσω να είμαι συντομότερη. Έχω να απαντήσω μερικά πράγματα για την ανεργία των νέων. Εάν εξετάσουμε τους αριθμούς, θα δούμε κάποια βελτίωση. Και αν κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ Απριλίου 2016 και Απριλίου 2015, θα δούμε ότι έχουμε 495.000 λιγότερους ανέργους. Λιγότερους ανέργους εν τέλει. Περί αυτό πρόκειται. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό, είναι καλή εξέλιξη. Βέβαια, μας μένουν 4,2 εκατομμύρια ακόμα. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένες με αυτή την εξέλιξη, όχι πάντως αρκετά. Και όταν εξετάζουμε τις ε, CSR, δεν τα λένε αυτά συνεχώς, τα λένε όμως στα εκτιμώντας. Δεν έχουμε ξεχάσει λοιπόν την ανεργία των νέων. Δεν έχουμε πατήσει το κουμπί που τη σβήνει. Ε, για μας είναι σημαντικό ακόμη διότι έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια νέους που ψάχνουν να βρουν δουλειά. Και ε, μπορώ να φανταστώ ότι είναι 4 εκατομμύρια ξεχωριστά ατομικά δράματα. Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν ότι όσο δεν έχουν προοπτική για δουλειά δεν μπορούν να αρχίσουν ε, μια οικογενειακή ζωή κλπ. Θα εφαρμοστεί τώρα η εγγύηση για τους νέους, θα δούμε ποια αποτελέσματα θα έχει. Έχουμε την προχρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή στήριξη. Είδαμε ότι βοηθεί στην χρηματοδότηση κάποιων έργων, κάποιων σχεδίων, κάποιων project από τα κάτω και θα επανέλθουμε. Αν χρειαστεί να δώσουμε περισσότερα χρήματα θα το ξαναδούμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση, mid-term review. Αλλά ας πούμε πάντως ότι οι διαθωτικές μεταρρυθμίσεις όντως λαμβάνουν χώρα. Υπάρχει μια μετάβαση στην αγορά εργασίας. Οι σχετικές υπηρεσίες λειτουργούν καλύτερα σε πολλές χώρες μέλη και δουλεύουμε πολύ σκληρά σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης, δηλαδή θέσεις εκπαιδευόμενων σε επιχειρήσεις ασκουμένων και ούτω καθεξής, με την βοήθεια βέβαια και των περιφερειακών αρχών, αλλά χρειάζεται να δημιουργηθούν οι θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται συνεργασία από πλευράς των επιχειρήσεων και να ενταχθούν στο ε, νέο ιδρυθέν αυτό σύμφωνο ε, υπέρ των νέων η πρόεδρος Λουσκόκ Ο κύριος Ουρτασούν για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Απευθύνω ερώτηση στον Αντιπρόεδρο κύριο Ντομπρόσκη σε σχέση με το Ισπανικό πακέτο. Στην σύστασή σας της 9ης Μαρτίου για την διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος λέτε ότι η μείωση του ελλείμματος ανακόπηκε από τις δημοσιονομικές συνέπειες της μεταρρύθμισης του ατομικού εισοδήματος. Δεν ξέρω, έχετε κάνει κανένα σχετικό υπολογισμό. Πρώτη μου ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτηση, στα πλαίσια πάντα της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, θέλω να ρωτήσω, κύριε Αντιπρόεδρε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ένα σενάριο όπου η Ισπανία συνεχίζει να μειώνει τους φόρους. Και θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο για ε, τέτοια μείωση. η κυρία Στάνοκα. Ευχαριστώ. Ερώτηση για τις ειδικέ συστάσεις ανά χώρα και τις κοινωνικές ε, συνέπειες τους. Εσείς, κύριε Ντομπρόσκης, είπατε ότι όταν κάνετε αυτές τις συστάσεις ε, δίνετε προτεραιότητα σε κοινωνικά και θέματα και θέματα απασχολήσεως. Έχετε ειδικά εργαλεία για να ελέγξετε πώς αυτές οι οικονομικές συστάσεις, πώς εφαρμόζονται αυτές οι οικονομικές συστάσεις. Και υπάρχει μηχανισμός για να γίνει το ίδιο και για τις συστάσεις που αναφέρονται στην απασχόληση. Την ίδια ερώτηση απευθύνω και στην Επίτροπο Τάισεν. Έχετε προτάσεις για το πώς μπορούμε να ελέγξουμε τι αποδίδουν οι, οι κοινωνικές ε, συστάσεις και αν εφαρμόζονται από τις χώρες μέλη. Και άλλη σχετική ερώτηση, τι να κάνει κανείς όταν ε, οι κοινωνικές συστάσεις έρχονται σε σύγκρουση με τις οικονομικές. Εσείς κύριε Ντομπρόφσκης, όταν ήσασταν Πρωθυπουργός της Λετωνίας το 2009, είχατε εισαγάγει μέτρα λιτότητας και από τα πρώτα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γνωρίζετε ότι τα μέτρα αυτά φύγουν ή έθιξαν τότε τα λιγότερο προστατευμένα στρώματα του λετωνικού πληθυσμού. Ευχαριστώ. Μάρκο Βάλι. Ευχαριστώ, παρεμβαίνω και εκπροσωπώντας άλλη συναδελφό μου. Για το ζήτημα της διακυβέρνησης, governance, η γραμμή της Κομισιόν είναι αρκετά σαφής. Βλέπουμε πώς λειτουργούν οι συστάσεις αυτές στην περίπτωση της Γαλλίας Και βεβαίω οι Γάλλοι πολίτε έχουν βγει στους δρόμους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Βλέπουμε παρόμοια πράγματα και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Η κερδοσκοπία έχει κυριαρχήσει παντού και η Κομισιόν ανοίγει τις πύλες για να ξεχυθεί η κερδοσκοπία και η κερδοσκόπηση ολόκληρη την Ευρώπη. Ακόμα και στις σημαίες, εθνικές σημαίες θα βάλουν το όνομά τους οι sponsors, οι διάφοροι χορηγοί. Αυτό το μέλλον φτιάχνεται για την Ευρώπη και συγχαρητήρια. Όπως είπε ένας Γερμανός συνάδελφος πριν, το ευρώ δεν αποδίδει, δεν λειτουργεί. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός Γερμανός που κατανοεί πραγματικά την κατάσταση, ότι το ευρώ, το οποίο μοιράζονται 19 χώρες, προκαλεί σημαντικές ανισότητες. Μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι στην ε, Γερμανία συγκεντρώνεται ένα σημαντικό πλεόνασμα, το οποίο θα μπορούσε να, να τοποθετηθεί σε φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης. και προτίθεστε να χρηματοδοτήσετε τις χώρες οι οποίες προβαίνουν σε μέτρα λιτότητας. τι; δύο λεπτά, ε, κύριε Σάντε. Μα έχω τρία λεπτά, κύριε. Ε, με ποιο δικαίωμα θα πείτε ότι δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο. Μήπως επειδή δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Έχω δύο σλότ από την πολιτική ομάδα, άλλα τρία λεπτά συνολικά. Η FTD είναι πολιτική ομάδα όπως και όλες οι άλλες. Γιατί δεν έχω τρία λεπτά. Ωραία, τα έχουμε γράψει σε βίντεο, αυτά τα στείλουμε σε όλη την Ιταλία να μεταδοθούν. Ε, ευχαριστώ. Ντόμινικ Μαχτά. Ευχαριστώ. Υπάρχει ο κίνδυνος επανάληψης. Θα ήθελα να σας ζητήσω αλλά μία ακόμη φορά θα πρέπει να πω άσχημα πράγματα, γιατί ασχολείται περισσότερα με τα ε, γεγονότα και λιγότερο με τις αιτίε. Πρέπει να υπάρξουν... Ε, ε λέτε ότι η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε και λέτε ότι πρέπει να συμμετέχουμε και έτσι δημιουργείται χώρες low cost. Ε, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην Ευρώπη. Αυτή η ελαστική ευελιξία, η κινητικότητα των εργαζομένων, η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, αγαθών, ε, αυτό σημαίνει ότι εκτός από την ανταγωνισμό που υπήρχε μεταξύ Βορρά και Νότου, υπάρχει και μια, ένας ανταγωνισμός Ανατολής και Δύσης που έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται θέσεις εργασίας και επομένω ανεργία. Επειδή Έχω μόνο 1,5 λεπτό. Δύο ερωτήσεις έχω να σας ε, θέσω. Πρώτον, για ποιο λόγο συνεχίζετε τις ε, διαπραγματεύσεις για το TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείες ενώ ε, η παραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών θα σκοτώσει την παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και παρά το γεγονός ότι έχουμε 25 εκατομμύρια νέους, 4 εκατομμύρια νέους, εξακολουθείτε να επιμένετε να υποδεχόμαστε ε, πολιτικούς και οικονομικούς πρόσφυγες, μετανάστες, διορθώνω, κάτι το οποίο θεωρείται ότι θα σημαίνει περισσότερα έσοδα για μας. Δίνω τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Ντομπρόφσκης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Για το πρώτο ερώτημα, τον προϋπολογισμό της ε, Ισπανίας και τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, για τον φόρο εισοδήματος. ο φόρος αυτός ε, προσωπικού εισοδήματος ε, είχε ως σκοπό να να αντισταθμιστεί από κάποια ισοδύναμα μέσα. Ε, μπορώ να σας δώσω λίγο περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, αλλά αυτή είναι η δική μας αξιολόγηση. Τώρα, κατά πόσο υπάρχει περιθώριο ελιγμών αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στην περίπτωση της Ισπανίας να μειώσει το χρέος της 3% ε, ε, του ΑΕΠ ε, και 2,5% το 2017. Αυτό βέβαια δυνάμει των αποφάσεων που θα ληφθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Συνεπώς, όσο η Ισπανία δίνει προτεραιότητα στις στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής της και αντισταθμιστικά ε, μέτρα. Στην προκειμένη περίπτωση μείωση του φόρου προσωπικού ε, εισοδήματος. Αυτό είναι δυνατό, δηλαδή δεν συζητούμε ε, με τόση λεπτομέρεια την κατάρτιση του προυπολογισμου εσοδα έσοδα-έξοδα. Είναι μια Συμβουλή Γενικής Πολιτικής ε, για τα κράτη-μέλη η φορολογία τους να περάσει από το χαμηλό μισθοεργατικό ε, δυναμικό ε, σε άλλους τομείς που είναι λιγότερο επιβλαβείς για την ανάπτυξη όπως η κατανάλωση, η ακίνητη περιουσία, πράσινη φορολόγηση κλπ. Εξαρτάται λοιπόν από την συνολική εικόνα και ο φόρος εισοδήματος είναι μόνο ένα τμήμα των στοιχείων αυτών. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα της ισορροπίας ε, ε, μεταξύ δημοσιονομικών, οικονομικών, χρηματοπιστωτικών έναντι οικονομικών, ενάντι κοινωνικών συγγνώμη, ε, στοιχείων που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι πράγματι κινούμαστε, κινούμαστε προς μια κατεύθυνση ώστε να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη ε, κοινωνικά κριτήρια, κάτι το οποίο συνέβη και στη Λετωνία, όταν έπρεπε να περάσουμε, να ολοκληρώσουμε ένα πρόγραμμα προσαρμογής πάρα πολύ δύσκολο, ε, με εισαγωγή ενός επιπλέον κοινωνικού δικτύου ασφαλείας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Όσον αφορά τώρα στο ερώτημα της γενικής ε, πολιτική, κατεύθυνσης πολιτικής ε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια ε, δημοσιονομική τάση που είναι αρκετά αυξητική σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ξέρω βέβαια ότι αυτή η ανάπτυξη δεν κατανέμεται ίσα μεταξύ των μελών της Ευρωζώνης και όσον αφορά το πλεόνασμα της Γερμανίας, πράγματι ε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τμήμα της σύστασής μας προς τη Γερμανία και γι' αυτό ακριβώς ε, η Γερμανία θεωρείται ε, ότι είναι χώρα στην οποία υπάρχουν οικονομικές ανισότητες και θα πρέπει το διαθέσιμο δημοσιονομικό του χώρο να το χρησιμοποιήσει για να ενθαρρύνει την επένδυση και την οικονομία. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ελεύθερης ε, κυκλοφορίας ε, αγαθών, ε, υπηρεσιών, προσώπων, Προφανώς ε, είναι οι ελευθερίες αυτές η βάση της ε, εσωτερικής αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς ε, είναι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτές τις τέσσερις ελευθερίες να τις υπερασπιστείς. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται και σχόλια σε περίπτωση καταχρήσεων. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την ΤΙΤΙ, πράγματι συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές. Είναι μία από τις ε, πρώτες προτεραιότητες διαπραγματεύσεις ε, σε εμπορικό επίπεδο και βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, απτά ε, αποτελέσματα εκατέρωθεν του Ατλαντικού για, αν ε, ε, υπάρξει συμφωνία για το TTIP. Τώρα όσον αφορά την προσφυγική κρίση, κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο θέμα, δεν είναι ακριβώς βέβαια το θέμα της δικής μας συζήτησης, αλλά πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να βοηθήσει ανθρώπους που χρειάζονται διεθνή προστασία. Και παράλληλα είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών, όπως επίσης και να ενισχύσουμε την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί βέβαια τμήμα της δουλειάς μας κατά την αντιμετώπιση της προσφυγικής αυτής κρίσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τάισαν πολύ σύντομα, γιατί ε, ο Βάλτης νομίζω απάντησε τις περισσότερες ε, ερωτήσεις, να απαντήσω όσον αφορά την ε, υποδοχή των προσφύγων, γιατί το κάνουμε και γιατί οργανωνόμαστε στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο θεωρούμε υπάρχει κάτι που το λέμε ηθική και συνείδηση, έχουμε μία νομική υποχρέωση αλλά και μία ηθική υποχρέωση να υποδεχθούμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πραγματικά αναζητούν προστασία για να μπορέσουν να σωθούν, να σωθεί η ζωή τους. Και Νομίζω ότι με 507 εκατομμύρια ε, πολίτες ε, νομίζω ότι μπορούμε να ε, φιλοξενήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζητούν βοήθεια. Το κάνουμε εμείς όπως το κάνει και πολλοί άλλος κόσμος σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να υποδεχθούμε το μερίδιό μας των ανθρώπων αυτών που αναζητούν τη βοήθειά μας. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν οι διεθνείς ε, συμφωνίες, αλλά και γιατί θέλουμε να βοήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Ήθελα να πω κάτι για το TTIP, αλλά νομίζω ότι ο Βάλτης ε, απάντησε, οπότε μπορώ να ολοκληρώσω εδώ, ε, κυρία Πρόεδρε, μήπως έτσι δώσουμε δυνατότητα να τεθούν περισσότερες ερωτήσεις. Περνάμε μόνο 1,5 λεπτό. Ο κ. Μοσκοβισή δεν είναι εδώ, οπότε θα κάνω ρωτήσεις στον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κάνετε συστάσεις για τη Γαλλία που δακτυλοδεικτούν ε, τις ε, αδυναμίες του φορολογικού μα συστήματος. Δεν βοηθάει την οικονομική ανάπτυξη, δεν ευνοεί τις παραγωγικές δυνάμεις και κυρίως λέτε ότι ευνοεί την κατανάλωση. Και επίση λέτε ότι είναι άκαμπτο ο γενικό δασμολογικό μα, ο γενικό φορολογικό μα κανόνα. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η φορολόγηση τη κατανάλωση μέσω αύξηση του ΦΠΑ και να καταργηθούν οι εξαιρέσει και οι χαμηλοί συντελεστέ. Αλλά είναι ακριβώ αντίθετο από αυτό που πρέπει, αυτό που λέτε. Πρέπει να μειώσουμε το ΦΠΑ και να μειώσουμε και αυτού οι οποίοι φορολογούνται. Τι στόχου έχετε η φορολογία είναι το τελευταίο προπήριο της εθνικής κυριαρχίας. Θέλουμε στη Γαλλία ένα σύστημα ενιαίο συντελεστή, όπως στις βαλτικές χώρες. Τέτοιες ε, φορολογίες είναι και κοινωνικά παράδεκτες, αλλά και οικονομικά αναποτελεσματικέ. Γιατί θέλετε να επιβάλλετε σε όλα τα κράτη-μέλη ένα μοντέλο. Αν η Κομισιόν θέλει να γίνει δημοφιλή, θα πρέπει να ασχοληθεί με το επίγον καθήκον της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών. Θα πρέπει, για παράδειγμα, οι τεχνολογικές επιχειρήσεις όπως η Google να πληρώνουν τους φόρους του στα κρατη Το θέμα αυτό είναι δική σας αρμοδιότητα. Οπότε, κύριε Ντομπροφσκής, σας ρωτώ, θα υπάρξει τελικά και μία φορολογική ένωση στην πράξη χωρίς να λέγεται στα λόγια? Λούντεκ Ευχαριστώ. Το πρωί ακούσαμε τον πρόεδρο του Eurogroup να μιλάει για την εφαρμογή των φορολογικών κανόνων. Επανερχόμεθα σε πρακτικές του παρελθόντος, για τις οποίες δεν είμαστε περήφανοι. Τώρα εξετάζουμε τις αναχώρα συστάσεις. Το 2012, 11% των συστάσεων ε, εφαρμόστηκαν 60% σε ένα βαθμό και 29% δεν εφαρμόστηκαν καθόλου. Τα τελευταία στοιχεία λένε ότι μόνο 4% έχουν εφαρμοστεί πλήρως, 44% εν μέρη και 52% καθόλου. Πιστεύουν λοιπόν οι επίτροποι ότι το σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο που καθορίστηκε πριν από λίγα χρόνια λειτουργεί και θέλω να σας θυμίσω ότι στόχο μας πρέπει να είναι να έχουμε υπεύθυνε πολιτικές, δεν είναι να έχουμε μια τέτοια ιδεολειπτική πολιτική. Δεύτερη ερώτηση. Δεν καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα. Λένε ότι θέλουμε να μειώσουμε τις συστάσεις ανά χώρα. Κοίταζα τι γίνεται στην Τσεχία. Και τι βλέπω. Αναφέρεστε στα ε, ευάλωτα παιδιά και τη συμμετοχή στην αγορά και την έρευνα και ανάπτυξη. Και επίσης βλέπω βλέπω ότι κάποιες παρόμοιες ε, συστάσεις ε, στο παρελθόν δεν έχουν εφαρμοστεί. Άρα τι έννοια έχει αυτή η μείωση. Ευχαριστώ. Ρωμάνα Τόμς. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, θετικό είναι το ότι λαμβάνουμε απευθείας απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Κανείς από εμά δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει, κανείς δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει μάλλον, ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο με ένα κοινωνικό μοντέλο που είναι επίσης το πιο ανεπτυγμένο. Αυτή η επιθυμία που έχει διατυπωθεί ο στόχος αναφέρεται σε πολλά κείμενα. Έχουμε ιδρύσει διάφορες υπηρεσίες για να εφαρμόσουμε αυτούς τους στόχους. Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι πολλοί από αυτούς τους στόχους ε, είναι μονολόγια. λόγια. Υπάρχουν σύμφωνα σταθερότητας, ε, υπάρχουν προγράμματα μεταρρυθμίσεων, αλλά δεν εφαρμόζονται. Πάντα όταν πρέπει οι δεσμεύσεις να εφαρμοστούν, ξαφνικά προκύπτουν ε, προβλήματα. Και δεν καταλαβαίνω, είναι θέματα τακτικής κάποιων αδύναμων κυβερνήσεων ή ήταν προγραμματισμένο κάτι τέτοιο. Το ίδιο ισχύει και για τη Σλοβενία. Οι μεταρρυθμίσεις που υποτίθεται ότι έπρεπε να εφαρμοστούν δεν εφαρμόζονται. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογή του. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξή. Εάν επιθυμούμε να αντιδράσουν τα κράτη-μέλη, όχι μόνο η δική μου χώρα, αλλά και τα άλλα κράτη-μέλη, εάν θέλουμε να εφαρμόσουν με πιο υπεύθυνο τρόπο τα κράτη της ε, συστάσει, πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνεται αν δεν τις εφαρμόζουν. Οπότε, η ερώτησή μου, έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε πίστα στα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τις συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης. Ευχαριστώ. για τις συστάσεις για την ε, φορολόγηση στη Γαλλία. Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, τη διαβάζω, να ληφθεί δράση για να, μειωθεί το χρόνο, το, να μειωθούν οι τάξεις οι φόροι στην παραγωγή, διευρύνοντας την ε, φορολογική βάση για την κατανάλωση, ιδιαίτερα όσον αφορά το ΦΠΑ, να καταργηθούν ε, οι μη αποτελεσματικές δαπάνες, ούτως ώστε οι φόροι οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα να καταργηθούν. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι συστάσεις μας δεν λένε ότι κάποιος φόρος πρέπει να είναι κλιμακωτός ε, ή με ένα μόνο συντελεστή. Οι συστάσεις είναι σύμφωνες με τις ε, γενικές αρχές για τη φορολογική πολιτική, για τις συμβουλές επιφορολογικής πολιτικής της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέμε ότι δεν πρέπει να φορολογείται η εργασία ιδιαίτερα χαμηλόμισθη, αλλά πρέπει να περάσει η φορολόγηση προς την κατανάλωση και αλλού. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν για τη Γαλλία είναι ε, σε γενικές γραμμές ε, σύμφωνο με αυτά που προτείνουμε και για άλλες χώρες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Γαλλίας. Τώρα τι κάνουμε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Το ανέφερα στις αγωγικές μου παρατηρήσεις η Επιτροπή θα κάνει μια σειρά από προτάσεις και έχει ήδη κάνει μια σειρά από προτάσεις και το θέμα αυτό είναι μία από τις κύριες προτεραιότητές μας. Τώρα, για το πώς εφαρμόζονται οι συστάσεις. Όντως και η Επιτροπή ανησυχεί. διότι για πολλές συστάσεις υπάρχει μόνο περιορισμένη πρόοδος. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε και να έχουμε καλύτερο διάλογο με τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η εφαρμογή. Αλλά και πάλι, παραλαμβάνω, δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής των ε, συστάσεων. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες μέσω της ε, μακροοικονομικής αιρεσιμότητας για τα προγράμματα επενδύσεων που μπορούν να βοηθήσουν ε, την εφαρμογή των συστάσεων. Αλλά πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι να επινοήσει ένα μηχανισμό κυρώσεων για την εφαρμογή των συστάσεων. Θεωρούμε ότι Αυτέ οι στάσει είναι προ το συμφέρον των κρατών μελών. Και τα επόμενα χρόνια θα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τη μέθοδο του καθορισμού τιμών αναφοράς όπως αναφέρει και η έκθεση των πέντε προέδρων το δεύτερο στάδιο συγκεκριμένα ούτως ώστε να είναι νομικά πιο δεσμευτική αυτή η χρήση τη μόνο αναφοράς. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται μάλλον ε, να συμφωνήσουν οι συνομοθέτες για το θέμα των συστάσεων γενικά. Ορισμένες φορές καλύπτουν πολλούς τομείς πολιτικής. Γι' αυτό θέλουμε να εστιάσουμε μέσω του εξαμήνου. Θέλουμε και λιγότερες λοιπόν συστάσεις που να καλύπτουν και λιγότερους τομείς πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπο Στάση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη για τις ε, συστάσεις αναχώρα, αν είναι λιγότερες ή περισσότερες. Για να απαντήσω τον κύριο Μαϊερ. αυτές έχουν ομαδοποιηθεί και από πριν οι συστάσεις δηλαδή και τώρα επίσης ομαδοποιούνται η πρόοδος στις χώρες μέλη σχετικά με τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Εμείς δεν βασιζόμαστε μονάχα στις εκθέσεις που μας υποβάλλουν οι χώρες μέλη, αλλά και στα στατιστικά δεδομένα για την ανεργία, την απασχόληση κλπ. Και έχουμε αναπτύξει δείκτες, έχουμε θεσπίσει δείκτες δηλαδή σε συνεργασία με τις χώρες μέλη για να μπορούμε να μετρούμε την πρόοδο που επιτελούν. Και χρησιμοποιούνται αυτοί οι δείκτες. Ο Βάλτης Πρόσκης αναφέρθηκε ήδη στην χρήση και των ε, ε, ταμείων και των μακροοικονομικών όρων. Και το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι όλο και περισσότερο στοχευμένες στα, σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία πρέπει να αποδεικνύονται. Και στηρίζουμε τις διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις, ώστε στο μέλλον να αναμένουμε πραγματικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε και εσείς κύριε Επίτροπε, ερώτηση όμως προς τον κύριο Ντομπρόφσκης. Αρχίζει να ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις διαστάσεις της ζώνης ευρώ, ιδίως με μια ετήσια παρουσίαση της ε, καταστάσεως. Πέραν όμως από την αρχική αυτή τοποθέτηση. Λαμβάνεται αυτό υπόψη στις αναχώρα συστάσεις, επειδή υπάρχουν βεβαίως και διασυνδέσεις μεταξύ των οικονομιών. Θέλω να έρθω τώρα στην διαδικασία για τις μακροοικονομικές ελλείψεις ισορροπιών. πέντε σοβαρά τη διαδικασία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην επιθυμία της να εφαρμόσει όλους τους κανόνες αυτό ο συγκεκριμένος κανόνας, τον οποίο έχει κρίνει και το παρόν Ευρωκοινοβούλιο, εφαρμόζεται και αν εφαρμόζεται πώς εξηγείται ότι οι χώρε που για πολλά χρόνια συνεχώς βρίσκονται πέραν των κατοφλίων που ρυθμίζει, που θεσπίζει η διαδικασία, δεν κάνουν τίποτε παραπάνω, δεν γίνεται τίποτε παραπάνω δηλαδή. Και δεν χρησιμοποιείται όλη η εργαλειοθήκη που προβλέπει νομοθεσία. Δεν λέω ότι πρέπει να επιβάλλονται κυρώσει σε όλο τον κόσμο, αλλά απλώς λέω, εφόσον υπάρχουν οι κανόνες, εγώ πάντως είχα κατανοήσει ότι οι κανόνες έχουν σκοπό να εφαρμόζονται. Ποια είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μόνο για ε, το έλλειμμα, αλλά για όλους τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Ευχαριστώ. και Λόπες, εσείς. Ευχαριστώ. Με εκπλήσει ότι υπάρχει τόσος εφησυχασμός στην ε, τοποθέτησή μας. Ενώ έχουμε τόσο υψηλή ανεργία, ενώ ο πληθωρισμός είναι γύρω στο μηδέν, ενώ οι ανισότητες ε, αποχαλινώνονται και η ανάπτυξη είναι ανεμική. Και τόσος κόσμος ε, ζει στα όρια της φτώχειας. Είναι σαφές ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι που καθορίσαμε και οι στόχοι για την αγορά εργασίας, δηλαδή η μείωση των αποδοχών και η ελαστικοποίηση των όρων εργασίας, οδήγησαν σε αποπληθωρισμό. Είναι τέταρτος χρόνος ε, τελικά στασιμότητας και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Παγκόσμια Τράπεζα. Βεβαίως ε, έγιναν δύο λάθη αύξησης των επιτοκίων εν μέσω κρίσης και όλα αυτά τα πληρώνουμε. Και όλα αυτά οδήγησαν σε ύφεση. Το πρόβλημα είναι ότι αν όλοι κάνουμε οικονομίες ε, την ίδια στιγμή, δεν αγοράζει κανείς, άρα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και αν περικόπτουμε τα εισοδήματα και τους μισθούς, ενώ κάποιοι διατηρούν τα προνόμια τους, θα το πληρώσουμε. Η επιθετική λοιπόν ε, δημοσιονομική εξυγίανση λειτουργεί, λέγεται, και τι γίνεται, ευελιξία για την αγορά εργασίας για να αντιμετωπιστεί η μείωση των εισοδημάτων. Δηλαδή, τι γίνεται στην Ισπανία. Έχουμε όλο και πιο επισφαλή συμβόλαια. Και σε τελευταία ανάλυση αυτό οδηγεί τελικά και σε μείωση των φόρων. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Ιβάνο Μαλέτη. Εσείς την εκπροσωπείτε. αντικαθιστώ τη συνάδελφο. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Τα σχόλια που έκανε ο Γερούν Ντάισεμπλουμ σήμερα το πρωί δείχνουν και πάλι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει τις, ε, τους κανόνες του MIB και δεν έγινε ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια δέσμη 6 μέτρων. Ίσως χρειαζόμαστε μια νέα δέσμη. Ε, μας είπατε ότι θα υποβάλλετε προτάσεις σε σχέση με την αύξηση της εθνικής κυριότητας των προγραμμάτων, περισσότερη, περισσότερος διάλογος και ελπίζουμε σύντομα τα εθνικά συμβούλια ανταγωνισμού σε όλα τα κράτη-μέλη αν δεν χρειαζόμαστε ένα πραγματικό καρότο, ένα πραγματικό κίνητρο προς τα κράτη-μέλη για να κάνουν κάτι, να συνδέσουν τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση με την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία ή στα ευρωομόλογα που θα μπορούσε να συνδέεται με αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφορετικά δεν μπορεί εκ των υστέρων να ζητήσει την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Τι είδου μείγμα μέτρων εκ των υστέρων και οικονομικών κινήτρων θεωρείτε ότι ότι έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τόμας Μαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ερώτηση προς την κυρία Τάισιν. Στις ε, συστάσεις αναχώρα λέτε ότι η ροή προσφύγων και μεταναστών έχει σημαντικές κοινωνικές συνέπειες και βραχυπρόθεσμα αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υψηλότερες δημόσιες δαπάνες και μεσοπρόθεσμα κάποια επιτυχία όταν θα έχουν ενσωματωθεί οι πρόσφυγε και οι μετανάστε. Συμφωνώ με αυτό. Στην Επιτροπή Απασχολήσεω είχαμε και έκθεση, εγώ ήμουν ο της του Λαϊκού Κόμματο, ακούσαμε πάρα πολύ διαφορετικές απόψεις, τελικώς καταφέραμε να συμβιβαστούμε. 36 συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες και τελικώ συμφωνήσαμε και υπερψηφίστηκε η έκθεση. Συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται διδασκαλία γλωσσών. Συμφωνήσαμε επίση ότι με κανένα τρόπο δεν πρέπει να μειωθεί ο κατώτατο μισθός ε, και για τους πρόσφυγες. Πρέπει να παραμείνει η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Είπαμε ότι θέλουμε αύξηση των πόρων των, του κοινωνικού ταμείου. Άλλοι ευρωβουλευτές είπαν ότι θέλουν και θέσπιση ειδικού ταμείου. Εμείς είπαμε ότι έχουμε το ΆΜΙΦ που είναι ένα ταμείο με πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση για πρόσφυγες μετανάστες κλπ. Και ότι θα ήταν εσφαλμένο το μήνυμα να έχουμε βραχυπρόθεσμα μεν υπέρ των προσφύγων πολλά χρήματα και για μεσοπρόθεσμα μέτρα σχεδόν τίποτα. Τι θα γίνει τελικά, θα συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πρώτα τους πόρους του ΑΜΙΦ ή θέλει τελικώς να φτιάξει ένα ειδικό ταμείο το οποίο θα έχει και ένα ειδικό δικό του τίτλο. Ευχαριστώ. Κύριος Μαριάς. Ήθελα να ρωτήσω, I would like to put a question for Mr. Dombrovski. Ε, ερώτηση για τον κύριο Dombrovski, αλλά θα, θα το πω στα ελληνικά. Ε, άκουσα τις προτάσεις σας και βλέπω ότι ακολουθείτε τον ίδιο δρόμο, δηλαδή την ίδια αποτυχημένη συνταγή. Να επενθυμίσω ότι έχουμε 40% του ελληνικού πληθυσμού που ζει κάτω από τα ωραία της φτώχειας. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Παρά τα αυτά με το τρίτο μνημόνιο επιβάλλονται και καινούργοι φόροι, που σημαίνει ότι διαλύεται η οικονομία. Ταυτόχρονα το τρίτο μνημόνιο απαιτεί αυξημένα πλεονάσματα της τάξης του 3-3,5%, πράγμα που σημαίνει ότι αφαιρεί πόρους από την ίδια την οικονομία. Το θέμα του χρέους επίσης δεν έχει ρυθμιστεί, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στο πώς θα λειτουργήσει η ίδια η οικονομία. Επομένω, μπαίνει ένα θέμα. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανέργους. Έχουμε σπάσει ρεκόρ στην ανεργία των νέων. Περνάει το 50%. Το ίδιο και στην ανεργία γενικότερα. Με ποια μέτρα λοιπόν θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα. Πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά. Διότι οι χιλιάδες νέοι ζητούν μία λύση. Περιμένουν να βρουν δουλειά. Και δεν άκουσα συγκεκριμένα μέτρα από τα οποία να προκύπτει πράγματι η δυνατότητα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν δουλειά. Διότι με τα μέτρα που προτείνεται, προφανώς σε 15 χρόνια να υπάρχει μια λύση. Αλλά τα χρόνια αυτά είναι πάρα πολλά για να μπορέσει να αναμείνει ο ελληνικός λαός αυτή την καταιγιστική πολιτική που επιβάλλεται με τη λιτότητα και τη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βάλε, θα έχετε τη δυνατότητα μία ακόμη φορά να θέσετε ένα ερώτημα παρά το γεγονός ότι ε, η πολιτική σας ομάδα δεν είχε αποφασίσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ναι, συγγνώμη για προηγουμένως. Νομίζω ότι υπήρξε μία παρεξήγηση με τη, μεταξύ της ομάδας μου και της γραμματείας. Λοιπόν, η συνάδελφος Σομπερές μίλησε για το πλεόνασμα. Δεν πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια ούτε για τη Γερμανία, ούτε για τη Γαλλία. Δεν ξέρω που είναι ο κύριος Μοσκοβισή, μπορεί να κρύβεται ξέρω εγώ, ίσως προσπαθεί να σχεδιάσει μια, την, την επόμενή του επίθεση σε μια άλλη χώρα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν έχουμε ένα κοινό νόμισμα πρέπει να υπάρχει και μηχανισμός αντιστάθμισης το οποίο να λειτουργεί. Οι χώρε με πλεόνασμα πρέπει να επενδύουν το πλεόνασμά του σε φτωχότερε χώρε. Διαφορετικά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να δούμε αυτή την ε, οικονομική νομισματική ένωση, γιατί όχι μόνο δημιουργεί ανισότητες, ανεργία και, και άλλα προβλήματα, διαφορετικά σε, μερικές, ε, σε μερικά χρόνια θα έχουμε ακόμη πιο καταστροφικές ε, καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς για για τις διαστάσεις της ε, Ευρωζώνης. Όντως, στη διάσταση μας της Ευρωζώνης. Ε, ε, πράγματι αποδίδουμε περισσότερη προσοχή τώρα και γι' αυτό προωθούμε και τη σύσταση για την Ευρωζώνη μαζί με την AGS, ώστε να επιτρέψουμε στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης όταν συντάσσουν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα να το αυτό υπόψη και αυτό απηχείται και στις αναχώρα συστάσεις που δίνουμε στις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η λογική πίσω από την αλλαγή αυτή στο εξάμεινο. Τώρα για τις μακροοικονομικές ανισότητες, τη σχετική διαδικασία δηλαδή. Συμφωνώ με την δήλωσή σας ότι οι κανόνες που υπάρχουν οφείλουν και να εφαρμόζονται και αυτό βεβαίως ε, οφείλει να ισχύει για όλους τους κανόνες. Τώρα, πιο ειδικά, για χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία έλλειψης ισορροπίας ή υπερβολικού ελλείμματος. Από φέτος έχουμε κάνει ένα streamlining στις κατηγορίες αυτές, στις διαδικασίες μακροοικονομικής αστάθειας και όλες οι σχετικές χώρες υφίσταται ειδική παρακολούθηση, ειδικό monitoring. Και όπως είπα, με περισσότερες και πιο εξειδικευμένες συστάσεις και με πρόσθετο monitoring σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους. Τώρα, για τις οικονομίες της Ευρωζώνης. Πράγματι υπάρχει οικονομική ανάκαμψη, πολύ μετριοπαθής όμως. Άρα, μέχρι 1,8% ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά για φέτος και οι προτεραιότητες μας είναι τα διευθυντικά ταμεία για να ενισχυθεί αυτή η ανάκαμψη. Και πάλι λέω για το ερώτημα όπως είπατε και εσείς την επιθετική φορολογική, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό βεβαίως χρειάζονται μέτρα που αυξάνεται. Ε, επίσης, σχετικά με τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε κίνητρα και αντικίνητρα και πώς να ενισχυθεί αυτή η ιδιοκτησία εντό εισαγωγικών των αναχώρα συστάσεων. Δηλαδή χρειάζεται οι εθνικοί φορείς, κυβερνήσεις, κοινοβούλια, κοινωνικοί εταίροι και στην περίπτωση των χωρών συνοχής και οι μακροοικονομικοί όροι, υπάρχουν και μακροοικονομικοί όροι, που μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των αναχώρα συστάσεων. Όμως η βελτίωση των αναχώρα συστάσεων και η εφαρμογή τους αποτελούν τον στόχο μας σε ό,τι αφορά και τις φετινές συστάσεις αλλά και για τον επόμενο κύκλο που αναζητούμε τρόπους για να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι συστάσεις αυτές. Τώρα, για το ερώτημα σχετικά με την Ελλάδα, για να είμαι σαφής, όταν συζητούμε τώρα το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τις αναχώρασεις τάση, η Ελλάδα δεν εντάσσεται σε αυτό το εγχείρημα, γιατί η, χώρα, η Ελλάδα ως χώρα προγράμματος δεν μπαίνει σε αυτό τον μηχανισμό παρακολουθήσης. Αλλά αυτά περιλαμβάνονται σε μνημόνιο κατανόησης. και τα έχουμε δει αυτά πρόσφατα. Το πρόγραμμα, είναι η αξιολόγηση έχει, έχει αξιολογηθεί, το πρόγραμμα προχωρεί, αναμένουμε ήδη από το δεύτερο εξάμεινο να υπάρξει ανάκαμψη στην Ελλάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρέος, γνωρίζουμε ότι η Ευρωομάδα, το Eurogroup, συμφώνησε να εγκύψει και στο θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και να λάβει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Και οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των εθνικών ελληνικών αρχών και τα τελευταία χρόνια και τώρα έχουν συμβάλει στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ώστε μπορούμε να αναμένουμε ότι η Ελλάδα θα επανέλθει στο δρόμο της ανάκαμψης και της δημιουργίας απασχόλησης που είναι τελικά και ο στόχος του προγράμματος και είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Τώρα για το ε, πλώνασμα των, των τρεχόντων ισοζυγίων στην Γερμανία. Η Γερμανία είναι σε διαδικασία πλεονασμάτων και αυτό που συστήνουμε στην Γερμανία και είναι η πρώτη μας σύσταση, νούμερο ένα σύσταση, ζητούμε επενδύσεις ιδίως σε υποδομές, σε καινοτομία και ανανέωση, να χρησιμοποιηθούν πόροι από το πλεόνασμα, να αντιμετωπιστούν προβλήματα υποχρηματοδότησης υποδομών και το καθεξής. Αυτό είναι το περιεχόμενο των συστάσεών μας προς την Γερμανία. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή το δημοσιονομικό περιθώριο που διαθέτει για να προσφέρει κίνητρα για ανάκαμψη. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Ουλφσκογκ. Κυρία Τάισεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω την ερώτηση του κυρίου Λόπες σε σχέση με τον κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας, ειδικότερα για την Ισπανία, γιατί το έχουμε θέσει αυτό το θέμα και στην έκθεση για την Ισπανία, αλλά στις αιτιολογικές σκέψεις, γιατί καταρχάς ε, θεωρήσαμε ε, ότι η Ισπανία ήταν μια χώρα στις οποίες υπήρχαν ε, κάποιες ε, ασυνήθιστες συμβάσεις εργασίας, περισσότερο από τις άλλες χώρες και γι' αυτό ζητήσαμε μεταρρυθμίσεις και ζητήσαμε και πληροφορίες για ε, την συνέχεια των μεταρρυθμίσεων αυτών για να ε, τα λάβουμε υπόψη ε, στις συστάσεις μας. Είδαμε βέβαια με χαρά ότι έγιναν κάποιες μεταρρυθμίσεις και είναι καλό που υπήρξαν αυτές. Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Μαν σε σχέση με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, κοιτάξτε, ε, ναι, στην αρχή θα υπάρχει ένα κόστος γιατί πρέπει να ενσωματωθεί ο κόσμος, έχουν τραύματα, έχουν προβλήματα, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της στέχασης, πρέπει να τους υποδεχθούμε, αλλά μετά υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μια ομαλή ε, και λειτουργούσα ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών όπως και με άλλους ε, ε, υπηκόους τρίτων χωρών που ζουν στις χώρες μας πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και πρέπει να τα κάνουμε και καλύτερα από ό,τι πριν γιατί όταν βλέπουμε πώς έχουμε ενσωματώσει ήδη υπάρχοντες υπηκόους τρίτων χωρών αν βλέπουμε για παράδειγμα τη στέγαση, την εκπαίδευση κλπ βλέπουμε ότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες ε, τώρα τις ε, αξιοποιούν, δεν τις έχουν. Είναι διαφορετική η κατάσταση για τα περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Και την περασμένη εβδομάδα υπήρξε και ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης για ε, υπηκόους τρίτων χωρών και για αυτούς που βρίσκονται εδώ αλλά και για αυτούς που μόλις έρχονται και για τους πρόσφυγες. Πρέπει λοιπόν σε πολλά επίπεδα να προσπαθήσουμε να τους ενσωματώσουμε και για την κοινωνία και για την κοινωνική συνοχή και για την οικονομία. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους ενσωματώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο το δυνατόν συντομότερα. Κατά πόσο έχουμε χρήματα. Υπάρχει υποστήριξη. Βρήκαμε. Βρήκαμε κάποια χρήματα 100.000 ε, μαθήματα γλώσσας θα γίνουν online ε, και πρέπει να χρηματοδοτηθούν, να χρηματοδοτηθούν. Βρέθηκαν τα χρήματα αυτά, αλλά πρέπει και τα κράτη-μέλη να ε, βάλουν και αυτά τον νοβολό τους. Όπως ξέρετε μπορούν να χρησιμοποιήσουν το FIRT e για τις πιο άμεσες ανάγκες, για να, για να καλύψουν τις πιο άμεσες ανάγκες, όπως και το EMSF για την το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για ε, την ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών και ε, για ε, μαθήματα γλώσσας κλπ. Όπως επίσης να υπάρξουν υπηρεσίες στις χώρες μέλη, όχι μόνο για να εξηγήσουν πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα, αλλά να υπάρξει και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γιατί τα κράτη-μέλη μπορούν να μάθουν από τις βέλτιστες αυτές πρακτικές και έτσι γίνονται τα πράγματα καλύτερα από το να πρέπει κανείς να τα κάνει όλα μόνος του. Ε, με την εξαίρεση των μαθημάτων αυτών εκμάθησης γλώσσας πρέπει να ζήσουμε με τον προπολογισμό που έχουμε στη διάθεσή μας βέβαια. Οπότε δεν ε, νομίζω ότι στο, κοινωνικό ταμείο, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα υπάρξουν περισσότερα χρήματα. Θα δούμε τι θα γίνει με την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να διαθέσουμε κάποια χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να ε, υποστηρίξουμε την ενσωμάτωση των ε, προσφύγων σε όλα τα κράτη-μέλη. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους για τις ε, παρεμβάσεις σας. Θέλουμε μια οικονομικώς αποδοτική Ευρώπη, αλλά θέλουμε αυτό να συμβεί και υπέρ της ε, απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ενός καλύτερου μέλλοντος για τους νέους ανθρώπους, ε, άνδρες και γυναίκες, όπως επίσης και για τους ηλικιωμένους. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Σίγουρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν όλους και καλό βράδυ.